Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στις ε, επεξηγήσεις ψήφου και θα ήθελα όλοι σας να φύγετε και να ακούσουμε αυτούς οι οποίοι πρέπει να λάβουν το λόγο ή που θέλουν ακόμα να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ αποχωρήστε ταχαίως ώστε να μπορέσουν να ομιλήσουν οι επεξηγούμενη. Ερχόμαστε λοιπόν στις εξηγήσεις ψήφου. Καταρχήν για το ψήφισμα για, την, ε, για τις εκπομπές των ελαφρών αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων. κύριο Μπένσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ επέλεξα το όχι στο μπλοκάρισμα των νέων κανόνων για τις εκπομπές από ελαφρά επιγατηγά και εμπορικά οχήματα που συμφώνησαν τα κράτη-μέλη και κομισιόν. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι εκπομπές ελέγχονται σε πραγματικές συνθήκες και όχι στο εργαστήριο. Αν είχαμε μπλοκάρει τους νέους κανόνες που είχε συμφωνήσει η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη, για πολλά χρόνια θα είχαμε ένα νομικό κενό χωρίς να ξέρουμε πότε θα έχουμε τις πραγματικές δοκιμές που θέλουμε. Θα ήταν σαν να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο με μια κουκούλα πάνω από τα μάτια, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι με τους νέους κανόνες δίνουμε επιταγή εν λευκό στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες στους οποίους ε, συμφωνήσαμε. Φυσικά θα πρέπει να προσαρμοστεί η βιομηχανία και θα πρέπει Εμεί να έχουμε φιλοδοξία για περιορισμό των εκπομπών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε σε μια ετήσια αναθεώρηση των εκπομπών και δεσμεύτηκε να μειώσει τις οριακές τιμές μέχρι το 2017. Ο κύριος Δεμεσμέκερ για ένα λεπτό. Οι εκπομπές, ειδικά τα οξύδια του αζότου, ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία. Σε ένα πανεπιστήμιο στις Ηνωμένε Πολιτείε έγιναν δοκιμές και είδαν ότι στο Βέλγιο έχουμε ειδικές, ειδικά προβλήματα με τον, την ποιότητα του αέρα και 1.200, 1.200 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ε, προσπαθούμε λοιπόν ε, στη Φλάνδρα με πράσινα οχήματα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για να περιορίσουμε τι εκπομπέ. Ακόμα υπάρχει μεγάλη ευελιξία, γιατί δεν έχουμε ακριβώ τι δοκιμέ ε, των εκπομπών σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Αυτέ οι δοκιμέ θα πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι απαράδεκτο να το δεσμεύσουμε αυτό με τα πρότυπα της Ευρώπης ε, Euro 6 που είναι χαλαρά και μιλάμε για 80 ε, μιλιγκράμμ το κιλό. Είναι σημαντικό αυτό ε, και πρέπει να το υποστηρίξουμε για λόγους υγείας. Ο κύριος Χάν για ένα λεπτό. Όλοι ξέρουμε ότι οι εκπομπές, ε, το σκάνδαλο των εκπομπών της Volkswagen ήταν σκάνδαλο. Υποτιμήσαμε ωστόσο πόσο καταστροφικό ήταν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν χωρίς λόγο λόγω μιας πολιτικής, της Ένωσης αποκλειστικά, μετά από το λόμπι των επιχειρήσεων. Από την Ένωση μόνο σε όλο τον κόσμο που προωθούσαν το δίζελ ε, που για πολλούς ήταν μέχρι τότε ήταν το κακό προϊόν. Οι Αμερικανοί άλλοι μιλούσαν για ευρυδικά αυτοκίνητα. Η Ένωση αποκλειστικά προώθησε την χρήση ενός καυσίνου που παράγει 40 φορές περισσότερα ε, νητρικά και 22 φορές περισσότερο ρηπογόνα ε, ε, σωματίδια. Δεν ξέρουμε πόσοι πέθαναν από καρκίνο, από καρδιά. Υπάρχουν ωστόσο χιλιάδες θύματα, θύματα των λόμπι των επιχειρήσεων και εμείς είμαστε όλοι ένοχοι, συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα. Ο κύριος Πίπερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σπάνια άκουσα να, λέει, να υπάρχει μια τέτοια κινδυνολογία όπως αυτή του προλαλήσοντος. Εγώ υποστήριξα την πρόταση της έκθεσης. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει πολύ ταχαίως μια πρόταση για να μπορέσει να εξασφαλίσει σταθερότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τους προμηθευτές της. Γι' αυτό καταψήφισα την ε, αίτηση καταψήφισης της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, κάλιο ένα και στο χέρι, δύο και καρτέρι. Αυτή ήταν η λογική μου. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε την ανασφάλεια σε σχέση με τον σχεδιασμό των προσπαθειών μας και επίσης έχουμε πετύχει και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε μια ευθύνη έναντι του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και των καταναλωτών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος και επίση ο κύριος Ζούντο Μπενίτο Σουλουάγα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς υπερψηφίσαμε της, ε, υπέρ της, ε, του εμποδισμού της μείωσης των, της, μάλλον της αποδυνάμωσης των ε, ορίων για τις εκπομπές γιατί υποστηρίζουμε τους πολίτες και όχι τις επιχειρήσεις. Το σκάνδαλο της Volkswagen γνωστό ως Dieselgate επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η πρόταση της Κομισιόν μονάχα εκπροσωπεί τη θέληση των ίδιων ατόμων που εδώ και πολλά χρόνια μας κορόιδευαν και μας εξαπατούσαν για τις εκπομπές θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα αυτού του τομέα. Εκατομμύρια θέσεις εργασία είναι αμφιβόλο και επίσης κινδυνεύει και η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών η ρήπανση από τα μικροσωματίδια και από τα οξύδια του αζότου οδηγεί σε μισό εκατομμύριο πρόοδους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε την μετακίνηση των επιχειρήσεων με το να έχουμε βιώσιμη οικολογικά και καινοτόμα αυτοκινητοβιομηχανία η οποία δεν εξαπατεί. Δεν πρέπει λοιπόν να δεχτούμε να καταπατώνται τα συμφέροντα όλων από τα συμφέροντα μοναχαρισμένων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλανκό Λόμπες για ένα λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, η έκδοση, η εκπομπή των ε, νετρικών υπερβαίνει πέντε φορές περισσότερο τα όρια. Ζητώ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αποσύρουν το κείμενο και να θα αυξάναμε ωστόσο, εάν δεν εγκρίναμε το κείμενο αυτό, την ασφάλεια δικαίου και θα, υπήρξε, και θα υπήρχε ε, σαφής βελτίωση της υγείας. Με το ψήφισμα, με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί κατά το ίμιση η εκπομπή και η Ευρώπη θα είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που έχει τόσο αυστηρές ε, ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Μόνο με την εφαρμογή των προτύπων αυτών θα τήρηθει η νομοθεσία, θα προστατευτεί το περιβάλλον, η υγεία, θα δοθούν εγγυήσεις στους καταναλωτές και χρήστες και θα παροτρύνουμε τις επενδύσεις και την απασχόληση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έναν τομέα που είναι πολύ σημαντικός για χώρες όπως ε, η Ισπανία, η δική μου. Ευχαριστώ. Γέζη Πόσπισε, λέει ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της αντίρρησης. Πιστεύω ότι οι κανόνες που προτείνει η Κομισιόν, που θα εφαρμοστούν από το 2017, είναι μια πραγματική και στεναρή βάση για δοκιμές σε συνθήκες πραγματικές οδήγησης. Στην Τσεχία ε, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ σημαντική και δίνει δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες Τσέχους. Θέλουμε σαφείς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμοστούν και για την αυτοκινητοβιομηχανία, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο για, τα, για τη συμπεριφορά των μεμονωμένων οχημάτων. Ψήφισα υπέρ της πρότασης Κομισιόν και η Κομισιόν ελπίζω να εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2017 όλο το σύστημα θα είναι λειτουργικό. Η κυρία Τόρες Μαρτίνες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς υπερψηφίσαμε την αντίρρηση αυτή γιατί το πιο απαράδεκτο από όλα είναι ότι η Κομισιόν θέλει να αποφασίσει χωρίς την διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, θέτοντας και πάλι σε κίνδυνο την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη. Το να διπλασιάσουμε τα όρια για τις εκπομπές διοξιδίων του αζότου είναι μια απαράδεκτη παραχώρηση στις μεγάλες πολιτικές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την περίπτωση της Volkswagen, όπου ήξερε η Κομισιόν ότι γινόταν αυτή η απάτη και παρόλα αυτά με την συνενοχή της συνέβαλε για να γίνει μια τεράστια απάτη των καταναλωτών. Θα πρέπει να, επα... να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιπτώσεων και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και διαφάνεια δεν είναι ένα απλό θέμα, ένα τετριμένο θέμα. Είναι θέμα της δικής μας ζωής και της ζωής των μελλοντικών γενεών σε αυτόν τον πλανήτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τακουλά για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σημαντικό το ότι ασχολούμεθα με το θέμα αυτό στην Ευρώπη και στην αυτοκινητομηχανία για να φτάσουμε στο σωστό όριο εκπομπών. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πέραν του περιβάλλοντος πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι αυτοκινητομηχανίες παγκόσμια θα πετύχουν χαμηλές εκπομπές. Η πρώτη της Επιτροπής είναι λοιπόν αποδεκτή αν προωθηθεί και νομίζω ότι βασικά στην Ευρώπη θα πρέπει να δούμε και τη δική μας ανταγωνιστικότητα και την, ε, τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με σεβασμό των ίδιων κανόνων. Το εμπόριο είναι παγκόσμιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ. <coughs> Κύριο Καπούτο, ένα λεπτό. Ψήφισα ε, κατά της αντίρρησης ε, για τα οχήματα ευρώ 6. Το Κοινοβούλιο δεν το δέχτηκε και δεν χάσαμε μια ευκαιρία για να συνταχθούμε υπέρ των πολιτών. Μετά το σκάνδαλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε την υποχρέωση να δώσει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες ούτω ώστε να έχουμε πιο βιώσιμε παραγωγέ οχημάτων. Δεν δεχόμαστε όρια εκπομπών πιο ψηλά από αυτά που ψηφίσαμε το 2007. Όταν ψηφίζουμε, δεν μπορούμε να θεωρούμε μόνο ε, να σκεφτόμαστε μόνο τα συμφέροντα της βιομηχανίας και όχι των πολιτών. Είμαστε εδώ κυρίως για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Οι πόλεις μας έχουν ε, φοβερό νέφο και ε, μονοξίδιο, διοξίδιο του αζότου, μικροσωματίδια που έχουν τεράστιο κόστος για την υγεία των πολιτών. Ζολταν Μπάλτσο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. την προηγούμενη δεκαετία υπήρξαν κάποιες θετικέ αλλαγές για την μείωση της ε, ρήπανσης του αέρα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Είναι μεγάλος ο αριθμός των προώρων θανάτων, μπορεί να φτάνει τις 400.000. Τα προβλήματα τα οποία είδαμε το φθινόπωρο του 2015 καταδεικνύουν ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν υπάρχει σεβασμός του νόμου. Το σκάνδαλο της Volkswagen κατέδειξε ότι χρειαζόμαστε να γίνουν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Η πράξη εφαρμογής της Κομισιόν δεν θα εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Με το να δεχτούμε αυτή την πρόταση, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2020 οι τιμές ε, οι οποίες έχουν προβλεφθεί μπορούν να, υπάρχει υπέρβασή τους κατά δύο φορές. Γι' αυτό το λόγο εγώ υποστήριξα την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίκη Πρόεδρος. Σόλο Λόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της αντίρρησης και είμαι ικανοποιημένη που απορρίφθηκε η αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο καονισμός της Κομισιόν θα είναι ενισχύ θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι μια καλή λύση. Ε, έχουμε αυστηρές οριακές τιμές και πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να τις εφαρμόσει και η αυτοκινητοβιομηχανία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι δοκιμές θα γίνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. και νόμιζα ότι είναι καλή λύση για τους παραγωγούς και για μας τους χρήστες που χρησιμοποιούμε διζελοκινητήρες. Οι αλλαγές στο καθεστώς των μετρήσεων είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση και πιστεύω και ότι, ότι και οι παράγοντες, η μόρφωση προτείνονται είναι καλή. Τέλος, ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως και οι συνάδελφοί μου στο Φιναγκάλ στο, στην ομάδα του ΕΛΚ, καταψήφισα αυτή την έκθεση. Νομίζουμε ότι έχει κάνει αρκετά η Κομισιόν. Μας αρέσουν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε σχέση με το σημείο αυτό. Αν προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της Κομισιόν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι θα έχουμε ένα πλαίσιο για πιο αποτελεσματική εποπτεία. Ε, θα γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία στα κράτη-μέλη, ανεξάρτητη διαδικασία ελέγχου επίση. Αυτή η πρόταση θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν να λάβουν δράση κατά ε, των τεχνικών υπηρεσιών που είναι πολύ χαλαρές ε, στην εφαρμογή των προϋποθέσεων έγκρισης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρος ερχόμαστε στην έκθεση Reading για τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Υπηρεσιών ΤΙΖΑ. Η κυρία Ντάρλιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με, την... με το ψήφισμα για τις διαπραγματεύσεις ΤΙΖΑ ζητούμε από την Επιτροπή να αλλάξει την πορεία στις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν υποστηρίξαμε τη συμφωνία ΤΙΖΑ. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία πρέπει να βοηθήσει, όχι να αποδυναμώσει την αναδιαμόρφωση του παγκοσμίου εμπορίου υπηρεσιών. Οι πολίτες έχουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η φωνή αυτή ε, είναι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικά Εκλεγμένο Κοινοβούλιο. Αντί να ασκούμε τις ευθύνες αυτές με ευθύνη ε, ε, σήμερα, κάποιοι ευρωβουλευτές προτίμησαν μια ανεύθυνη στάση μόνο και μόνο για να βγουν στον τύπο. Πρέπει να υποστηρίξουμε το δίκαιο εμπόριο και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στην σχετική μας δράση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και η ομάδα μου καταψήφισα το ψήφισμα για ένα βασικό λόγο αυτό που θέλει να επιτευχθεί μέσω της συμφωνία ΤΙΖΑ είναι η μετατροπή σε αντικείμενο κέρδους και εμπορικό αντικείμενο βασικές θεμελιακές ε, δράσεις του κράτους, την υγεία, την παιδεία. Εμείς πιστεύουμε ότι η κοινή διαχείριση των ε, κοινών αγαθών πρέπει να είναι στο κέντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες TTIP, TISA κλπ προχωρούν μια διαδικασία απορρίθμισης εις βάρος της κυριαρχίας των πολιτών που δεν ενημερώνονται και βλέπουν σταυριακά να τους αφαιρούνται κομμάτι αποφάσεων του μέλλοντος τους. Καταψηφίσαμε το TTIP και την TISA, ζητούμε να ακουστεί η φωνή εκατομμυρίων πολιτών που είναι αντίθετοι με αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος Χένον έχει το λόγο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συχνά κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για το βρετανικό δημοψήφισμα μας λένε η συμμετοχή της Ένωση είναι αναγκαία για τις υπηρεσίε. Ωστόσο εμεί είμαστε εδώ συζητώντα μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της υπηρεσίες που περιλαμβάνει πέραν της Ένωσης άλλα 22 κράτη του ΟΣΑ από το Περού μέχρι την Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά κράτη ε, της Ένωσης δεν μετέχουν γιατί στην ουσία εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις αυτές μόνο με την Επιτροπή. Για χώρες που έχουν μεγάλη εμπλοκή στον τομέα των υπηρεσιών αυτό είναι κακό. Μπορεί να πετύχουμε πολλά πράγματα στον κόσμο αν μπορέσουμε να ξαναδούμε τη θέση μας στον κόσμο σαν μια ναυτική δύναμη με μεγάλη εμπορική παρουσία. Η κυρία Μακοβέη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σήμερα υπερψήφισα τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις της ΤΙΖΑ. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι μοναδική στην ιστορία λόγω της εμβέλειάς της, λόγω του περιεχομένου της και το ευρύ φάσμα θεμάτων που εμπλέκει. Χώρες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να συνεργαστούν σε αυτό το πλαίσιο. Προτείνει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μεγαλύτερες δράσεις και να μπορούν αυτές οι εταιρείε να αναλάβουν δημόσιες προμήθειες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε τρίτες χώρες και επίσης οι καλύτεροι επαγγελματίες να μπορούν να εργαστούν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι και τμήμα αυτής της πρότασης. Αλλά προφανώς κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την δική του ε, παρουσία στην αγορά υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεγκίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συνθήκη ΤΙΖΑ για τις υπηρεσίες είναι ένα καλό βήμα και χάρη στα Wikileaks ε, είδαμε λίγα από τα μυστικά έγγραφα και από τα λίγα που είδαμε ε, βλέπουμε ότι θα φύγει η ουδετερότητα του δικτύου ε, και πολλές άλλες κακές εκπλήξεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε διάφοροι. Δουλέψαμε σκληρά για το κείμενο που ψηφίσαμε σήμερα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξή ότι η υπογραφή της ΤΙΖΑ είναι μακρινή και η κίνηση Cinque Stelle ε, δεν είπε ναι στο ΤΙΖΑ, αλλά σε κάποιο είδους εντολή για τους διαπραγματευτές του ΤΙΖΑ που θα λέει ε, ξεκάθαρα ότι δεν αγγίζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν ε, μία αντιστρέψιμα και θα πρέπει τα συμφέροντα των πολιτών να πρετανεύουν σε σχέση με τις ελεύθερες συναλλαγές. Το κείμενο δεν είναι τέλειο, αλλά είναι σημαντικό να με αφήσουμε λευκή κάρτα στου διαπραγματευτέ, γιατί θα, κάνουμε, θα υποκληθούμε στα λόμπι θα είμαστε εμείς ε, άγρυπνοι γιατί καμία συνθήκη δεν ε, έχει πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τους πολίτες. Τάκουλα ε, για ένα λεπτό. Τάκουλα, ένα λεπτό. ευχαριστώ. Η συμφωνία ΤΙΣΑ αναθεωρεί τη συμφωνία ΓΚΑΤ και αν κοιτάξετε το κείμενο οι δημόσιες υπηρεσίες αποκλείονται. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίζουν ποιες υπηρεσίες είναι δημόσιες ε, και η εκπαίδευση και η υγεία είναι εκτός του ΤΙΖΑ. Αναφέρθηκε ότι διαπραγματευόμαστε με άλλες 22 ε, χώρες όπως Αυστραλία, ε, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, άλλες και άλλες χώρες, 22 χώρες συνολικά του ΠΟΕ. Ε, το εμπόριο υπηρεσιών επεκτείνεται και σε αυτές τις χώρες που είναι φυσικοί εταίροι και αλλού. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό θα αυξήσει τι θέσει απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη και αν κατάλαβα καλά, το Κοινοβούλιο θέλει αυτή την ανάπτυξη στην Ευρώπη, θέλει περισσότερε θέσει απασχόληση και αυτό είναι ένα τρόπο, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο μέλλον. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, διάκοψα. Αλλά βάλαμε ε, καθυστερημένα το ρολόι και σας διάκοψα νωρίτερα. Ο επόμενος ομιλητής, ο Νικολά Καπούτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ που Υπερψήφισα την έκθεση διότι η ΤΙΖΑ είναι μια ευκαιρία για να απαγιωθεί η θέση της Ένωσης ως μεγαλύτερη εξαγωγή υπηρεσιών στον κόσμο αφού εδώ καλύπτεται το 70% του εργαζομένων στην Ένωση και το 40% των εξαγωγών της Ευρώπης. Η συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, διευκολύνοντας την διευθυνοποίηση των ΜΜΕ και ε, μειώνοντας τις μη δασμολογικές και δασμολογικές ε, παρεμβάσεις που πλήττουν τον τομέα. Είναι στρατηγική σημασία η πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά σε μια εποχή ψηφιακής οικονομίας που μέσω της ΤΙΣΑ μπορεί να γίνει και που που δίνουν μια δυνατότητα πρόσβαση. Κατά συνέπεια, η σωστή εφαρμογή των γενικών αρχών τη εμπορική πολιτική, θα ενισχύσει την ε, δυνατότητα τη Ένωση να κάνει την ΤΙΖΑ μια πραγματική πολυμερή ε, συμφωνία. Ε, η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την δημιουργία μια πιο ενοποιημένη αγορά υπηρεσιών που θα μειώνει το κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ και θα σέβεται το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάμικινς. μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η συμφωνία Τίζα είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την απελευθέρωση και φιλελευθερωποιεί σε διάφορους τομείς, μεταφορές, τράπεζες κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες προωθούν τη συμφωνία αυτή που θα έπρεπε να καλύψει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη. Θέλω να τονίσω την ανάγκη να αποκλείσουμε τις πολιτιστικές και οπτικοακουστικές υπηρεσίες από την ΤΙΖΑ για να κρατήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιάς στις νέες χώρες. Εν γέννη είμαι θετική. ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για το εμπόριο υπηρεσιών καλύπτει πολυμερείς συμφωνίες θέτει όμως σε κίνδυνο τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις υπηρεσίες θέτει ένα αμφιβόλο την απασχόληση, τις θέσεις απασχόλησης, τις δημόσιες υπηρεσίες και επίσης την κυριαρχική ικανότητα των κρατών μελών να ρυθμίζει αυτές τις υπηρεσίες. Είναι ένα βήμα ακόμα για την παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό το απορρίπτω. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ανοίγουν νέες αγορές για τις πολιτικές σε βάρος των πιο αδύναμων χωρών, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, θα πρέπει αντίθετα να προστατεύσουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις απασχόλησής τους και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να παρέχουν τα δικά τους αγαθά και τις δικές του υπηρεσίες και να απεφευθεί το ντάμπινγκ. Γι' αυτό κατεψήφισα. Ο κύριος Πόλτσακ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εντυπωσιάζομαι με τον τρόπο με τον οποίο πολλοί από τους συναδέλφους μου καταφέρνουν να μιλήσουν σε ένα λεπτό αλλά μετά φεύγουν χωρίς να ακούσουν τους υπολείπους. Δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία με το να φτιάνει τείχη γύρω από τα, την επικράτειά της θα αυξήσουν την ε, ευμαρία τους. 40% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ έχει να κάνει με υπηρεσίες διαμεθοριακού χαρακτήρα. Η φιλελευθεροποίηση έχουν <clears throat> εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευμάρεια σε όλους και θα επιτύχουν και σε αυτήν την περίπτωση να έχουν μεγαλύτερη απασχόληση όλοι. Θα πρέπει να φιλελευθερωποιήσουμε περισσότερο και να προστατεύσουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Τις ε, υπηρεσίες γενικού συμφέροντος τις έχουμε εξαιρέσει από τη Συμφωνία ΤΙΣΑ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε. Είναι απαραίτητο για μένα οι Δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις να μην τύχουν διακρίσεων εναντίον τους. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Σον Κέλλη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Υψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, όπως και οι συναδελφοί μου. όπως και άλλοι 531 ευρωβουλευτές, είναι μια μεγάλη πλειοψηφία που κέρδισε η Vivian Redding, η συνάδελφός μου, που έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Και με αυτές τις προτάσεις ε, θα έχουμε ευρύτερο εμπόριο στις υπηρεσίες ε, μεταξύ περισσότερων εταίρων και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Ε, είμαστε ο μεγαλύτερος ε, εισαγωγέας και εξαγωγέας υπηρεσιών και μπορούμε να υποφεληθούμε πάρα πολύ από την υποστήριξη και την οικοδόμηση ενός ε, αυστηρού και στεναρού κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς υπηρεσίες. Είναι πολύ σαφές λοιπόν ότι αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν την υλοποίηση αυτού του στόχου και θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο θέμα για επεξήγηση ψήφου που είναι το ψήφισμα για μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά μόνο μετά το 2015. Η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά υποστηρίξαμε αυτό το ψήφισμα, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Κοινοβούλιο ε, το είχε ζητήσει, την είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2011 είχαμε σαφώς επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική για την ε, ισότητα των γυναικών μετά το 2015. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εφαρμογή, σε όλο και πιο έντονη εφαρμογή των πολιτικών ε, φύλου και θα πρέπει ε, αυτή η πολιτική ε, για το φύλλο να διαπνέει όλες τις πολιτικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν καταφέρουμε την, ε, την ιδέα των ε, ίσων δικαιωμάτων των γυναικών να τη βάλουμε στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να κινούμαστε σωστή ατραπό. Ο επόμενος είναι η Μικέλα Τζουφρίντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών ε, έληξε το 2011. Όλα αυτά που έκανε ε, η Κομισιόν για το 2016 είναι ένα έγγραφο εργασίας για την ισότητα των φύλων για το 2016-19. Ποιος θέλει, όποιος θέλει να είναι κακόπιστος μπορεί να πει ότι πέρα από μια τόσο αδύναμη έτσι πράξη ε, και μια αποδυναμωμένη ανακοίνωση είναι η πολιτική έλλειψη θέλησης Κομισιόν να ασχοληθεί με το θέμα ισότητα. Έχουμε σαφέστατη ανισότητα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες και μητέρε και εργαζόμενες μητέρε οι γυναίκες. Ε, είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ε, φραγμούς που πρέπει να σπάσουμε. Δεν είναι ιδεολογία αυτά, είναι πραγματική ζωή. Ε, θα πρέπει να έχουμε διαφορά στους μισθούς, ε, μητρικές άδειες. Ε, νομίζω ότι η ισότητα των γυναικών είναι θέμα ε, πολιτισμού. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από, την από εργασία της Κομισιόν. Ελπίζω η Κομισιόν να κάνει κάτι παραπάνω. Το ελπίζω και το εύχομαι. Ο επόμενος... Ο κύριος Χάναν δεν είναι παρόν. Επομένως δίνω το λόγο στην Τάνια Γκονσάλες Πένιας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή μας παρουσίασε ένα κείμενο εργασίας, όχι μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Δεν περιλαμβάνονται στόχοι, προπολογισμό, δείκτες μέτρησης ή μεταγενέστερης αξιολόγησης. Η πρόταση της Επιτροπής αγνοεί το ψήφισμα του Ιουνίου του 2015 του Κοινοβουλίου και όχι μόνο, αλλά και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του ίδιου έτους. Ταυτόχρονα προϋποθέτει και ενδεχομένως μια υποχώρηση στο δρόμο για την ισότητα. Η Επιτροπή λέει ότι η ισότητα φύλων έχει πολιτική υποστήριξη. Τα γεγονότα ωστόσο δείχνουν πως πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Παραμένουμε στην πατριαρχική αντιμετώπιση. Ο αγώνας για την ισότητα των ανδρών με, τους, με, με τις γυναίκες πρέπει να είναι στο κέντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υπερψηφίσαμε το κοινό ψήφισμα που κατατέθηκε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκοβέη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Υποστήριξα την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2010-2015 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα καταψήφισα το ψήφισμα αυτό. Όχι γιατί είμαι αντίθετος με την ισότητα των φίλων, αλλά διότι δεν θέλω, θεωρώ ανεπαρκές να υιοθετούμε τη μία, το ένα ψήφισμα πίσω από το άλλο, που ουδέποτε υλοποιούνται και εφαρμόζονται. Γυρίζουμε στην πατρίδα μας και λέμε ψηφίσαμε και ένα ψήφισμα για την ισότητα των φίλων δεν λέμε όμως ότι δεν θα το εφαρμόσουμε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται η υλοποίηση των ψηφισμάτων και ας σταματήσουμε να εγκρίνουμε ψηφίσματα που είναι περιτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίτση, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Κομισιόν Μάλλον δεν χαίρομαι για το γεγονό ότι η Κομισιόν αγνώρισε το Κοινοβουλίο και δεν υιοθέτησε μια <clears throat> πολιτική για ενημερωμένη αντιμετώπιση των ε, διαφορών ανδρών και γυναικών. Το έγγραφο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και δεν υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο. Επομένως δεν θα μπορέσει να έχει τη σωστή προσέγγιση. Ο ρόλος μου σε Ω βουλευτού είναι να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική η οποία θα έχει μια πιο μακρόπνοα αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων και παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. Εγώ υποστήριξα λοιπόν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων που ζητά μια μεταρρύθμιση της στρατηγικής της Κομισιόν ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών, να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες πρόσβασής τους σε υψηλές θέσεις, όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιούρι Πόσπιλ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν υπεστήριξα το ψήφισμα σήμερα για την νέα στρατηγική που παρουσιάστηκε από την αριστερά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω όμως να ε, νομιστεί ότι είμαι εναντίον της ισότητας των φίλων. Εγώ την υποστηρίζω αυτή την ισότητα των γυναικών με τους άνδρες. Το θέμα είναι με ποια μέσα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Αυτά τα οποία παρουσιάζονται από την αριστερά πτέρυγα του Κοινοβουλίου δεν είναι καθόλου ε, λυσιτελή και δεν είναι και εφικτά. Τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα αποδεχτούν. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο του εφικτού και όχι των ευσεβών πόθων και των ασκήσεων επιχάρτου. Εγώ ενδιαφέρομαι λοιπόν να δω τι μπορεί να επιτευχθεί οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες παραδείγματος χάρη σε μεγάλες επιχείρησεις. Αυτό δεν ήταν επιτυχές. Ευχαριστώ. Άντες Μάνικινς, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, συμφωνώ με την πλειοψηφία των ε, Ευρωβουλευτών που θέλουν μια νέα στρατηγική μετά το 2015 για το θέμα αυτό. Ζητάμε επίσης από την Κομισιόν να ετοιμάσει ένα πραγματικό έγγραφο, όχι ένα έγγραφο εργασία απλώ. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τι αρχέ που χρησιμοποιούσαμε σε προηγούμενα κείμενα και στη νέα στρατηγική για μετά το 2015 και να εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ όχι μόνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και μεταξύ άλλων φορέων. Η προθεσμία θα πρέπει να είναι το 2020 δε, της στρατηγικής αυτής. Παρότι θα εντάσσεται στη νέα εκλογική, στη νέα περίοδο του Κοινοβουλίου, δηλαδή στη νέα κοινοβουλευτική θητεία, παρόλα αυτά πρέπει να υποστηρίξουμε το 2020. Ο Γιουρέκ, κύριος Γιουρέκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λάβαμε ένα νέο εγγραφό για την ισότητα των φύλων που βασίζεται σε μια ομφαλοσκοπική έτσι, αντίληψη που έχουμε. Μετά από τόσα χρόνια ε, θεωρούμε ότι η κοινωνική θέση της γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη. Όχι, στην πραγματικότητα ε, υποσκάπτουμε την σημασία του γάμου. Ε, υποτιμούμε επίσης τη σημασία των γονέων μέσα στην οικογένεια. Επίσης προωθούμε τις ε, αμβλώσεις που τις θέλουν και εύποροι άνδρες. Αυτή είναι η κατάσταση της γυναίκας. Αυτή είναι η σωστή θέση της. Όχι, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό. Θα πρέπει να κάνουμε αναστροφή, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε τη ζωή στην Ευρώπη. Να υπάρχει ζωή στην Ευρώπη. Λοιπόν. Δηλαδή. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα όπου εκφράζει την άποψή του για τη στρατηγική της Κομισιόν στον τομέα της ισότητας των φύλων. Ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι πραγματικά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα που κάνει έκκληση για μια νέα στρατηγική από τη Σύνοδο Κορυφής, αντί να υιοθετήσει ένα κείμενο το οποίο θα εστιάζει σε συγκεκριμένα βήματα, τα οποία πραγματικά θα βελτιώσουν τη θέση της γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της κυρίας Γιούροβα και μέσω αυτού του εγγράφου που μας παρουσίασε η Κομισιόν, αφορούν την βελτίωση της, θέ, της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα, ε, ίσους μισθούς, ε, ίσες συντάξεις, καλύτερη εκπροσώπηση στα δουσού των εταιριών και σε ιδιωτικές εταιρείε και σε δημόσιους φορείς. Αντί για αυτά, τι κάναμε, υιοθετήσαμε μια δήλωση που δεν λύνει τίποτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα για μένα να μπορέσω να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η προλαλή σας, γιατί για πολύ καιρό εγώ σκέφτηκα πώς θα έπρεπε να ψηφίσω σε σχέση με το ψήφισμα αυτό. Δεν βλέπω κανένα λόγο να μην υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα. Είμαι υπέρ της ε, αρχής ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών. Για μένα λοιπόν αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η ισότητα να αποτελεί μια βασική αρχή σε όλα τα συνταγματικά έγγραφα, σε όλες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα που είχαμε ενώπιόν μας έχει ζητήσει την πρόοδο σε τομείς όπως η βία κατά των γυναικών, ισότητα στον χρόνο εργασίας, την παιδεία, στην ε, περίταλψη. Όλα αυτά είναι θεμητά. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα και τελικά το υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο Σον Κέλλη. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Όχι ίστατος όμως. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι βασική αξία της Ένωσης. Και τα κράτη-μέλη, η Ιρλανδία μεταξύ αυτών, έχουν αναλάβει σημαντικά βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Υπήρξε ωστόσο επιβράδυνση τη πολιτική δράση και των ρυθμίσεων σε επίπεδο ένωση την τελευταία δεκαετία. Στην Ιρλανδία, παρά την πρόοδο, κάποια πρόοδο στον τομέα αυτό, υπάρχουν ακόμα σημαντικέ διαφορέ στου τομεί στου οποίου μετέχουν άνδρες και γυναίκες και η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα υψηλά επίπεδα. Ακόμα και σε κλάδους ε, όπου υπάρχει σημαντικά υψηλότερος αριθμός γυναικών, δεν ακούν τα πράγματα. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή τη νέα στρατηγική που ζητά από τα κρατη να λάβουν βήματα για την αντιμετώπιση των θεμάτων ισότητας και να εξασφαλίσουν την ίση της ισότητας ευκαιριών στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Έχουμε εκλογές ε, στην Ιρλανδία τώρα και 30% των υποψηφίων πρέπει να είναι γυναίκες. Αυτό είναι ένα καλό βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση και τις επεξηγήσεις ψήφου. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα.